Ευχαριστώ πολύ κύριε Καμπαντά. Παναγιά μου. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Α, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία 20 χρόνια ε, ο χώρος Σέγγεν έχει χρησιμοποιήσει τα ίδια τις ε, ίδιες θεωρήσεις ε, και ε, τώρα έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την τροποποίηση το, του μορφότυπου των θεωρήσεων. λόγω του ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, προτείνω να μην υποβάλουμε τροποποιήσεις. Πρόκειται για ένα μορφότυπο που έχει ήδη υποβληθεί στο ενδιαφερόμενα μέρη, έχουν ήδη προσαρμοστεί τα μηχανήματα ανάγνωσης και επομένως η νέα νομοθεσία θα πρέπει οπωσδήποτε το ταχύτερο να εγκριθεί λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα επίγωσα κατάσταση. Εάν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να υποβάλει τροπολογίες πάντως θα πρέπει να το κάνει μέχρι την 9 Δεκεμβρίου έτσι ώστε τον Ιανουάριο να προχωρήσει το θέμα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Παρεμβάσεις θέλει κάποιος το λόγο. Κύριε... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια πάρα πολύ καθαρή περίπτωση ο κύριος συνάδελφος Ζαμπάσκη ε, πραγματικά μας ε, το παρουσίασε πολύ απλά ε, είναι απαραίτητο να ξεκινήσει άμεση δράση έτσι ώστε να εκλείψει η πιθανότητα παραχάραξης ή απάτης. Υπάρχει άλλωστε και στην ε, νέα οδηγία ε, ε, μια νέα πρόβλεψη όσον αφορά την ισχύ και τη διάρκεια ισχύως του στίκερ. Όμως δεν αναφέρεται συγκεκριμένα το πώς ακριβώς μετριούνται οι έξι μήνες ε, και οι έξι μήνες ε, βάσει της οποίας θα πρέπει να γίνει ε, να ισχύσει η αυτοκόλλητη αυτή η ετικέτα θεώρηση το στίκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζευκά. Ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Έχουμε εκπρόσωπο της Κομισιόν και αν θέλει να πάρει το λόγο, όχι. Επομένως ε, υπενθυμίζω υποβολή τροπολογιών μέχρι την 9η Δεκεμβρίου και σας ευχαριστώ πολύ ε, κύριε συνάδελφε. Περνάμε στο σημείο 22. Ο κύριος Γκασμπάρα έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Ενημερωθήκαμε ότι ο εισηγητής ανέβαλε την παρουσίαση και την πήγε 23 Δευτέρου. Οπότε και σας ε, προτείνω να προσαρμόσουμε το θέμα των εργασιών μας ανάλογα με αυτή το διακανονισμό. Οπότε περιμένουμε την εισήγηση για το θέμα αυτό. Αυτό σας προτείνω. Και η παρουσίαση των ε, τροπολογίων και η συζήτηση να πάνε επομένως τέλη Φεβρουαρίου, αρχάς Μαρτίου. Πολύ καλή ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου. Αλλά δεν σα λέω γιατί. Ah Παρατηρήσει, euh, <laughs> Ωραία. Και πάμε στο επόμενο σημείο. Το 24. Madame Delvaux. Κυρία Ντελβό, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας πω τι γίνεται στον αφορά την ρομποτική και επίσης τις ε, ηθικές επιπτώσεις της ρομποτικής. Και όλα αυτά υπό την άγρυπνη υποπτία του κ. Άντερσον που είναι τακτικό μέλος αυτής μας της ομάδας εργασίας γιατί κάναμε μια συνάντηση και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται τι γίνεται με τη ρομποτική περίπλοκα τα πράγματα και πολύμορφα οπότε πάμε πρώτα για τον ορισμό του ρομπότ καταρχήν πρόκειται για βοήθημα υλικό που έχει ε, μηχανικό κομμάτι, ηλεκτρικό κομμάτι και μετά κάποιους άλλους ε, δέκτες και αισθητήρε και επίσης ε, συζητήσαμε το κατά πόσο να έχουμε ένα πρόγραμμα, έναν αλγόριθμο που ας πούμε να επεξεργάζεται τα του χρηματιστηρίου είναι αυτό ρομπότ και είπαμε ότι αυτό παίζεται, είναι αμφίβολο οι ε, εφαρμογές μπορούν να είναι επικύλες, παραδοσιακά έχουμε τα ρομπότ στην ε, βιομηχανία. Ήταν η πρώτη γενιά. Στο μεταξύ όμως είναι σημαντικό να μην ξεχνούμε ότι η Ευρώπη είναι ο πρώτος παραγωγός στον κόσμο για βιομηχανικά ρομπότ. Έχουμε 40% της αγοράς για τα ρομπότ των υπηρεσιών. Άρα είναι θέμα και βιομηχανίας για την Ευρώπη συχνά. Πάντω, τα ρομπότα ασχολούνται με κάποιε εργασίες ε, πολύ επικίνδυνες, ας πούμε υγιέ, φωτιές. Ε, Υποβρύχες εργασίες. Η Γεωργία χρησιμοποιεί πολλά ρομπότ. και υπάρχει ένας ε, τομέας με τα προσθετικά μέλη. Με αυτά τα πρόσθετα μέλη βοηθούν ε, τα ρομπότ. Επίσης θα ανοίξει μια μεγάλη αγορά με τα ρομπότ που θα βοηθούν τους ε, ηλικιωμένους ούτως ώστε να είναι πιο αυτοεξυπηρετούμενοι κάθε μέρα και επίσης κάτι που όλοι θα γνωρίζετε είναι τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό αλλά και τα αεροπλάνα χωρίς πιλότο. Για τα drones έχει κάνει ήδη η Επιτροπή Πολυμεθυρών μια έκθεση με συστάσεις Καλά να μην επικεντρωθούμε σε αυτό, αλλά πάντως ε, πέρσι τέτοια αεροπλάνα και αεροπλανάκια ήταν το πιο συχνό δώρο τα Χριστούγεννα υπάρχουν παντού όλων των ε, μεγεθών και δεν διέπονται από νομοθεσία και εν πάση περιπτώσει ό,τι υπάρχει δεν είναι ομοιογενές. Μπορεί να περάσει τα σύνορα έναν ντρόν χωρίς να το καταλάβουν και αν διαφέρει η νομοθεσία, η ασφάλεια και όλα αυτά από το ένα κράτος στο άλλο, ε, αυτό είναι πρόβλημα. Με όλα αυτά ασχολήθηκαμε και ανακαλύψαμε, τουλάχιστον για μένα έναν κόσμο δεν ξέραμε ότι υπήρχε Βέβαια το θέμα είναι το ηθικό ζήτημα. Νομίζω ότι είναι εύκολο να πούμε ότι θέλουμε να υπάρχει ένα κώδικα διοντολογία από κάποια επιτροπή για να καταλήξουμε σε κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ και να έχουν οι ερευνητέ που ασχολούνται με τα ρομπότ ένα τέτοιο κώδικα. Το θέμα είναι βέβαια αν όλοι έχουν του ίδιου ηθικού κανόνε. Όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε με εμπειρογνώμονες. Θα νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια πλαισίωση για πλευρά της ηθικής, από πλευράς. πολλά ερωτήματα. τι είναι ρομπότ, δεν είναι αποκλειστικά ρομπότ, είναι θέμα προστασίας ιδιωτικού βίου, το ρομπότ δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν υπάρξει κάποια ροή δεδομένων και φαντάζεστε να υπάρχει ένα ρομπότ με κάποιον ηλικιωμένο στο σπίτι του και θα πρέπει να έχει πληροφορίε για όλα όσα γίνονται στο σπίτι. Οπότε το ρομπότ έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και στο πώς διαχειριστεί Άρα το θέμα της προστασίας ιδιωτικού βίου είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Άρα βέβαια είναι ευρύτερο. Δεν είναι μόνο για τα ρομπότ, έχουμε την επιτήρηση, τις κάμερες, όλα αυτά. Οπότε γίνεται κουβέντα για το τελικό μπορεί να υπάρχει ένα κουμπί στο μπουτόν τόσο ώστε να απενεργοποιήσει τη ροή των δεδομένων. Να όπως και τα ε, αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Όλα θα πρέπει να έχουν ένα μαύρο κουτί, να καταγράφεται ό,τι γίνεται στο αυτοκίνητο στην περίπτωση ατυχήματος. Και αυτό το κουμπί off, αν υπάρχει, τι γίνεται σε περίπτωση ατυχήματος, τι γίνεται με την ασφάλεια. Είναι μπλεγμένα τα πράγματα τώρα. Δεύτερη πτυχή σημαντική για να μπορούν τα ρομπότ να ε, δουλέψουν είναι τα cyborg και τα δίκτυα ασφαλείας. Εκεί δεν υπάρχει πιστοποίηση για τα ρομπότ στην Ευρώπη. Ας πούμε ξαφνικά ενώ μιλάω κόβεται το κινητό μου. Αν αυτό συμβεί σε ένα ρομπότ στο δρόμο, τι θα γίνει. Πώς θα οδηγήσει κανείς αν δεν έχει τα δεδομένα. Όλα αυτά είναι μπερδεμένα και θα πρέπει να τα διερευνήσουμε. Αλλά δεν είναι οπωσδήποτε δουλειά της δικής μας Επιτροπής. Έχουμε στην ομάδα εργασία προσώπους άλλων επιτροπών. Άλλο τώρα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Το θέμα της ευθύνης. Ποιος έχει την ευθύνη αν υπάρξει με ένα ρομπότ ατύχημα, οι κατασκευαστές, οι χρήστες, το ίδιο το ρομπότ. Γιατί υπάρχει μια θεωρία στην Γαλλία ότι θα πρέπει να το αποδοθεί η νομική προσωπικότητα του ρομπότ. Ούτω ώστε ακριβώ το ρομπότ να φέρει την ευθύνη. Άρα, με θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Άλλο θέμα ελεπτυχή είναι αυτό το δικαίωμα για τη σύμβαση. Το δίκαιο των συμβάσεων. Τι γίνεται, γίνεται με τη συντήρηση, γίνεται με τις υπηρεσίες. Άρα θα πρέπει στη δική μας επιτροπή να το κανονίσουμε, να γίνει μια δηλαδή ακρόαση με εμπειρογνώμονες, διότι δεν συμφωνούν οι εμπειρογνώμονες. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση μεταξύ αυτών που είναι υπέρ της στενής αντίληψης της ευθύνης και αυτών που θέλουν να εξηγηθεί περιπτωσιολογικά και εκείνοι που θέλουν να έχει νομική προσωπικότητα το ρομπότ. Εγώ σηκώνω τα χέρια. Οπότε μοιράζομαι μαζί σας τις απορίες μου. Άρα, ζητώ από την Επιτροπή μας να το οργανώσει. Έχουμε εμπειρογνώμονες, αλλά θα ήταν ε, ενδιαφέρον να μπορέσουμε να αντιπαραβάλλουμε τις απόψεις επίσης. Υπάρχει και το ζήτημα των δικαιωμάτων του δημιουργού τι θα γίνει εάν κάτι δημιουργήσει το ρομπότ Πύριος έχει τα δικαιώματα επί αυτού του δημιουργήματος και αυτό να μας απασχολήσει. Ε, επίσης έχουμε θέματα ασφάλειας των εργαζομένων. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η πρώτη γενιά των ρομπότ στην βιομηχανία διεκνόντουσαν από σαφή διάκριση ανθρώπων ρομπότ και δεν ήταν σε επαφή γιατί πολλές φορές ε, ήταν πολύ επικίνδυνα τα ρομπότ και άρα ε, δεν γινόταν επαφή ανθρώπων ρομπότ αλλά όμως η δεύτερη γενιά στηρίζεται στην συνεργασία ρομπότ ανθρώπων άρα θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι κανόνες ασφαλείας στην εργασία ε, επίσης είναι το θέμα ασφάλειας για τους καταναλωτές πολύ σημαντικό και αυτό Επίση, υγεία. Πολλά ρομπότ στον τομέα τη υγεία. Χειρουργική. Καλύπτονται από τι ιατρικές συσκευέ, Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει αρκετός έλεγχο και <laughs> επαρκή πιστοποίηση. Και επίσης όλα τα ε, συστήματα για τα προστατά μέλη τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο. Επομένω, και εδώ μπαίνει θέμα ηθικής. Τι γίνεται, ο ρόλος είναι η, η βοήθεια όταν υπάρχει κάποια αναπηρία ή ο ρόλος του ρομπότ είναι να βελτιώσουν τον άνθρωπο με προσθετά μέλη, με βοήθεια και χωρίς να υπάρχει πρόβλημα υγείας και έτσι να μπορούμε να βελτιώσουμε, να ομορφύνουμε τέλο πάντων τον άνθρωπο. Ηθικά θέματα αναδύονται εδώ, τα οποία θα πρέπει βεβαίω να τα συμπληρώσουμε με τους ειδικού τα θέματα ηθικής. Νομίζω ότι ολοκλήρωσα για το θέμα αυτό και βέβαια ευχαριστώ πολύ την ΣΤΟΑ της Επιρεσίας έρευνας του Κοινοβουλίου. Κάναμε μια μελέτη για τα διάφορα σενάρια. Τι μπορεί να συμβεί στην επόμενη 20 ετία. Άρα περιμένω τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης ε, Φεβρουάριο, Μάρτιο θα προκύψουν. Και εγώ προτίθεμαι να έχω έτοιμη την εκθεσή μου τον Μάιο και έτσι όλοι θα μπορέσουν να τα αφομοιώσουν και στις άλλες επιτροπές και να γνωμοδοτήσουν. Πάντως αυτά τα οποία έμαθα από αυτόν τον ε, αξιοθαύμαστο ψημονικό κόσμο της ρομποτικής είναι ότι υπάρχει υπόθεση με πολύ μεγάλη ε, φιλολογία επιστημονική φαντασίας αλλά γίνονται και πράγματα, πραγματοποιούνται, οπότε θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι στην νομοθεσία και να μην φρενάρουμε την έρευνα και τις εξελίξεις. Να ξέρουμε όμως ότι οι αναπτύξεις είναι καταιγιστικές και άρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Δεν μπορούμε να παγώσουμε την εξέλιξη. Πρώτα πρώτα είχαμε τις μηχανές, στη δεύτερη γενιά είπαμε ότι χρειαζόμαστε τους κανόνες και στη συνέχεια ε, μιλάμε για 20-25 χρόνια για μια γενιά ρομπότ. Θα τα κάνουν όλα στη θέση των ανθρώπων. Να το μέλλον αυτών των αναβαθμισμένων, βελτιωμένων ανθρωπίνων όντων. Άρα να μην βιαστούμε, να νομολογούμε, να νομοθετούμε, να το συζητούμε, χωρίς να θεωρούμε ότι αύριο το ρομπό θα στραφούν εναντίον μας και θα μας αντικαταστήσουν σε όλα. Βέβαια είναι θέμα απασχόλησης, γιατί είχαμε εκείνη την συνάντηση που αφορούσε την απασχόληση. Οπότε σε αυτό το μέτωπο δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει, διχάζονται οι ειδικοί είναι κάποιοι που λένε ότι θα καλύψουν 60% των θέσεων εργασία, αλλά δεν λάβαν υπόψη ποιε θα είναι οι νέε δουλειέ. Βέβαια θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της εκπαίδευσης και της παιδείας, γιατί χρειάζονται άλλες δεξιότητες διαφορετικές από αυτά που θέλουμε σήμερα. Κατάρτιση, εκπαίδευση, σόβια, διαβίου κλπ. Άρα πρέπει κανείς και μια και δυο και τρεις φορές να εκπαιδεύεται για να προσαρμόζεται σαν εργαζόμενος στις εξελίξεις. Επίσης, να σας τονίσω ότι η Επιτροπή Απασχόληση έχει μια τέτοια ομάδα εργασίας. Ακριβώς για να ασχοληθεί ε, με την σχέση απασχόλησης και ρομποτικής. Δουλεύουμε λοιπόν από κοινού για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν ε, εμπειρογνώμονες ε, οι οποίοι λένε ότι υπάρχουν περισσότερο, ότι, ε, ε, ότι ε, χρησιμοποιηθούν περισσότερα ρομπότ στις, στην βιομηχανία, τότε η ανταγωνιστικότητα θα αυξηθεί και ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ξαναεπιστρέψουμε, στις, να, επιτρέψουμε τον επαναπατρισμό διαφόρων βιομηχανιών στην Ευρώπη και στις χώρες μας. Πάντως, βλέποντας τι συμβαίνει στις άλλες υπήρους, διαπιστώνουμε ότι και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ε, ε, χρησιμοποιούν μαζικά τη ρομποτική και η Κίνα επίσης έκανε τεράστιες επενδύσεις προς την ίδια κατεύθυνση, άρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποφύγουμε. Άρα καλύτερα είναι να προλάβουμε την κατάσταση και όχι να ακολουθούμε μόνο τα ρομπότ των άλλων χωρών. Αυτά ήθελα να σας πω. Βέβαια θα μπορούσα να μιλάω επί ώρες για το θέμα αυτό γιατί το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον και με παθιάζει αλλά εν πάση περιπτώσει να σταματήσω. Και θα ήθελα άμεσα να σας ζητήσω να διοργανώσετε ένα hearing, μια δημόσια ακρόαση ε, για τον νόμο, τον, το δίκαιο των συμβάσεων. Ε, ναι, ναι, καταλαβαίνω, λέει ε, ο πρόεδρος, καταλαβαίνω τον προβληματισμό σας. Ναι, βεβαίως, ε, φαντάζομαι, θα, θα ρωτήσουμε και τους συναδέλφους, αλλά νομίζω ότι όλοι θέλουν να μάθουν περισσότερα γι' αυτό. Μάλιστα, στο Βέλγιο υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι εμπειρογνώμονας, ο κύριος Λωρό Αλεξάνδρα, ο οποίος προέρχεται από τον ιατρικό τομέα, έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο που ονομάζεται «Ο θάνατος του θανάτου» ε, ε, και ναι, ακριβώς αναφέρει εκεί πώς ε, οι αλγόριθμοι αλλάζουν ε, με πολύ ουσιαστικό τρόπο την ε, ιατρική. Έχει ασχοληθεί επίσης με την ρομποτική στη χειρουργική. Στο Στρασβούργο μάλιστα, εδώ και τέσσερα χρόνια, γίνονται καρδιαγγειακές επε επεμβάσεις οι οποίες ε, γίνονται με μετάδοση από μακριά δεδομένων μέσω δορυφόρου ε, και αυτό είναι πραγματικά κάτι καταπληκτικό. Ο κύριος Άντερσον θέλει μήπως να πάρει το λόγο. Well, thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τον κύριο Ντελβό είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομάδα εργασίας. Είναι ευρύτατο το πεδίο και συναρπαστικό. Και έχει γίνει μεγάλη πρόοδος, πολύ περισσότερη από ό,τι πίστευα. Το μέλλον είναι πραγματικότητα πλέον. Και βλέπουμε ήδη πως πάρα πολλά πράγματα από αυτά που φανταζόμασταν θα γίνουν πολύ σύντομα. Αυτές οι εξελίξεις είναι ταχύτατες στη ρομποτική. Και βλέπουμε επίσης πως σε κάποιους τομείς οι εξελίξεις θα λάβουν χώρα είτε είμαστε εκεί είτε όχι. Γι' αυτό χρειάζεται νομοθεσία. Για παράδειγμα, Μία τέτοια περίπτωση είναι τα μη επανδρομένα μεν οχήματα, τα drones. Ήδη βρίσκονται στην παραγωγή, υπάρχει, ε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου συγκρούνται, εξαφανίζονται και πρέπει να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε ένα αριθμιστικό πλαίσιο για αυτά τα οχήματα. Υπάρχει επίσης ο τομέας ε, της τεχνητής νοημοσύνης, της ε, χειρουργικής με τη βοήθεια ρομποτικής και άλλοι τομείς. Τα αυτοκίνητα. Εάν όμως θέλουμε και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε εξίσου γρήγορες εξελίξεις και να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τότε πιστεύω πως ε, έχουμε ε, την ευκαιρία και μεγάλο δυναμικό κιόλα για πολιτική δράση, για να κάνουμε ε, τη διαφορά. Ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης πιστεύω πως θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ σημαντικά ερωτήματα τις ερχόμενες δεκαετίες. Γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε να ε, τις τα εξετάζουμε για να δώσουμε απαντήσεις από τώρα. Σίγουρα δεν περιμένω να βρούμε όλες τις απαντήσεις και να τις συμπεριλάβουμε στην έκθεση, όμως ίσως μπορέσουμε να βρούμε κάποιες από τις ερωτήσεις και αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο, κύριε Ζήπκα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι συναρπαστικό θέμα αυτό, πραγματικά. Δεν ήξερα πολλά γι' αυτό και σας ζηλεύω, οφείλω να ομολογήσω, κυρία εισηγήτρια, διότι μαθαίνετε τόσα πολλά για αυτό το πράγμα και πιστεύω πραγματικά πως μία ακρόαση θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη. Θα είχαμε τότε την ευκαιρία να μάθουμε πολλά και περιτώ να πω ότι προσπαθώ να θυμηθώ πώς ε, ήταν ένας υπολογιστής πριν 30 χρόνια και πώς ήταν η ζωή μας χωρίς το διαδίκτυο, ε, είναι ε, πολύ περίεργο. Και φανταστείτε τι θα γίνει σε 30 χρόνια από τώρα. Ο κόσμος της ρομποτικής θα είναι τελείως διαφορετικός. Υπολογιστές. 30 χρόνια νωρίτερα δεν κάναμε τις σωστές ερωτήσεις. Και οι εξελίξεις έγιναν ταχύτατα, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζαμε και από ε, την δυνατότητα που είχαμε να αντιδράσουμε. Και τώρα λοιπόν τα ρομπότ έχουν τη δική τους θέση στον κόσμο μας και χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλούς ε, τομείς. Εμάς μας απασχολούν ε, κάποιοι από αυτούς τους τομείς, η ασφάλεια, η ευθύνη, οι νομοθετικές ρυθμίσεις, δεν μπορώ να φανταστώ ένα ρομπότ να είναι μια νομική οντότητα, ένα νομικό πρόσωπο. Τώρα βέβαια, αλλά ποιο ξέρει πώς θα είναι τα πράγματα στο μέλλον. Στηρίζω επομένως απόλυτα την ιδέα που είχατε για να διοργανώσουμε μία ακόμα ακρόαση. Πρέπει να μάθουμε περισσότερα, πρέπει να δούμε τι μας περιμένει στο μέλλον. Και μπορώ να φανταστώ επομένως μία έκθεση τον Φεβρουάριο, μία κρόαση τον Μάρτιο και ολομέλεια ίσως τον Μάιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντελβό για αυτήν την έκθεση που μας κάνατε, παρουσίαση που μας κάνατε που ήταν και παθιασμένη και ευχάριστη. Το θέμα της ευθύνης ε, των ε, πραγμάτων ε, και η ιδέα της αντικειμενικής ευθύνης άνευ πτέσματος, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα επανέλθουμε στο ερώτημα, τα ρομπότ έχουν άραγε ψυχή ή όχι θα προσφύγουμε στις ε, μεγάλες ε, φιλοσοφικές ε, συζητήσεις και τις μεγάλες περιχριστιανισμού και ψυχής συζητήσεις έτσι ώστε να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά. Ωστόσο, εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία αφορούν, αφορούν μονάχα την καθημερινή μας ζωή. Αναφερθήκατε προηγουμένως στα αυτοκίνητα, αλλά ξέρετε, τα αεροπλάνα ήδη ε, λειτουργούν ήδη λέω με συστήματα ρομποτικής και μόνο και τα λίγα ε, δυστυχήματα που γίνονται τα αεροπορικά οφείλονται κατά κανόνα σε λάθη πιλότων και όχι σε λάθη μηχανών. Ε, όσον αφορά τη δεοντολογία τώρα και την ηθική, όταν ήμουν ακόμα νέος είχα διαβάσει ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας στο Βαμπότ όπου τα ρομπότ είχαν συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Ε, η, δεύτερη, η πρώτη ήταν να προστατέψουν ε, την πόλη και το δεύτερο, η δεύτερη υποχρέωση ήταν ότι έπρεπε να σώσουν ε, και να προστατεύουν τον κατασκευαστή τους. Αλλά βλέπουμε στο βιβλίο ότι εκρήγνεται τελικά το ρομπότ γιατί έπρεπε για να προστατέψει τον κατασκευαστή να σκοτώσει κάποιον. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το ηθικό ζήτημα. Τώρα, ε, η, ιδέα ότι οι πιο υποτιμητικές ή πιο δύσκολες δουλειές ε, δεν θα γίνονται πλέον από τους ανθρώπους αλλά από τις μηχανές ε, είναι ένα σημαντικό θέμα. Μπορεί κανείς να πάει στην Ιαπωνία ή στην Κίνα για να δει πώς υποκαθίσταται ο άνθρωπος σε πολλές περιπτώσεις από το ρομπότ. Αλλά το θέμα της φορολογίας ε, είναι ε, ένα θέμα ε, πολύ σημαντικό. Η δικιά μας η λειτουργία, η κοινωνία λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή από την μία πλευρά δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να φορολογήσουμε το εισόδημα έτσι όπως φορολο... τη μηχανή δηλαδή να τη φορολογήσουμε όπως φορολογούμε τον άνθρωπο αλλά ταυτόχρονα θα βρεθούμε απέναντι σε μεγάλη ανεργία. Όταν ε, ε, ε, βρισκόμαστε ας πούμε σε ένα hearing, σε μια ακρόαση και θέτουμε το ερώτημα, το ζήτημα της ρομποτικής, δεν θα πρέπει το ερώτημα να αφορά μονάχα την τεχνική πλευρά, τα τεχνικά σκέλη, αλλά και τα κοινωνικά και τα εργασιακά και τα φορολογικά. Ευχαριστώ. Έχετε πολλές ερωτήσεις. Α, όχι, δεν έχετε άλλες ερωτήσεις. Εγώ θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια ερώτηση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι παθιασμένο και σημαντικό. Και εγώ ως ε, ε, νεόφυτος το παρακολουθώ. Όταν θα έχουμε βρει, ας πούμε, τον υπολογιστή που θα είναι 15.000 φορές ε, πιο δυνατός από το από, τον παρόντα ε, υπολογιστή, αριθμομηχανή, τότε θα είμαστε σίγουρα σε θέση να γνωρίζουμε την φύση των ε, ε, όλων των στοιχείων θα ξέρουμε τα πάντα για τα μηνοξέα και τον τρόπο που λειτουργούν στον οργανισμό μας θα ξέρουμε ναι, 15.000 φορές δυνατότερους ε, αριθμομηχανές, κομπιουτεράκια, τότε θα πρέπει να περιμένουμε περίπου 20 χρόνια νομίζω. Οι τομείς που πρέπει να μελετήσουμε ε, αφορούν όλα αυτά τα οποία είπατε και τους τομείς που και εσείς αναφέρατε, όχι μονάχα τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της έρευνας στην Ευρώπη, γιατί χρειαζόμαστε κάποιες δημόσιες πλατφόρμες, όχι μονάχα και φυσικά όλο το κοινωνικό περιβάλλον και το νομικό περιβάλλον, που θα πρέπει να ε, υπηρετήσει την ουδετερότητα των ρομπότ όπως και την ουδετερότητα του ίντερνετ αλλά βεβαίως και όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν και σχετίζονται με την με την ε, δυνατότητα που θα έχουμε να ε, μελετήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια ακρόαση οπωσδήποτε προς τα τέλη του πρώτου τριμήνου ίσως και δεύτερο. Ε, φοβάμαι ότι θα είναι πολύ σύντομο το διάστημα. Θα πρέπει να ζητήσουμε όμως από τους εμπειρογνώμους, λέει η κυρία Ντελβό, να έρθουν αρκετά γρήγορα. Οι προσκλήσεις να φύγουν γρήγορα. Ναι, μπορούμε να κάνουμε πολλές ε, ακροάσεις γιατί είναι πολλά τα ζητήματα. Θα πρέπει οι συντονιστές να συμφωνήσουν από πού θα ξεκινήσουμε γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε σε μία ακρόαση και σε μία μέρα ε, να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα. Ούτε ή άλλως και εγώ προσωπικά τουλάχιστον μετά από τρεις ώρες δεν, ε, το μυαλό μου δεν μπορεί να, ακολουθεί, να παρακολουθήσει πλέον πιο περίπλοκα θέματα και περίπλοκες τοποθετήσεις οπότε καλύτερα θα ήταν περισσότερες παρουσιάσεις, να σχολιάσω. Συμφωνώ με τον κύριο Άντερσον. Δεν θα βρούμε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Ωστόσο, είναι καλό να τεθούν τα ερωτήματα, γιατί θα πρέπει να γίνει συζήτηση, όχι μονάχα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στην κοινωνία γενικά. Πού θέλουμε να πάμε, τι μας περιμένει, πώς θα τα οργανώσουμε όλα αυτά, πώς θα ε, οργανώσουμε την κοινωνική συμβίωση. Είναι φιλοσοφικό το ερώτημα και σίγουρα ξεπερνάει τον ακαδημαϊκό κόσμο ή κάποιους εμπειρογνώμονες ή ερευνητές θα μπορούσαμε να συζητούμε επί ώρες ε, για να αποφασίσουμε αν κάποτε θα αποκτήσουν ψυχή ή όχι τα ρομπότ. Δεν το ξέρω και για την ώρα κανείς δεν το ξέρει. Αλλά σίγουρα ε, είναι πραγματικά ένα μαγικό θέμα για όλους. Γιατί αυτή η προσήλωση στα ρομπότ ε, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει από την αρχαιότητα. Εγώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή απέναντι σε μια βεβαιότητα του τύπου «Μα θα βρούμε λύση για όλα, θα τα κανονίσουμε όλα, θα τα ρυθμίσουμε όλα». Εγώ θα ήθελα μια πιο συγκεκριμένη προσέγγιση, δηλαδή να πούμε τι μπορούμε να ρυθμίσουμε στην αρχή. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις. Ας πούμε, τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό είναι κάτι το οποίο πολύ σύντομα θα προκύψει και δεν θα είναι το Google Car γιατί θα σας πω τι έμαθα, ότι τα Google Cards μπορούν να λειτουργήσουν μονάχα όταν, ε, όταν έχει ήλιο και όταν τα αυτοκίνητα ε, ε, βρίσκονται σε κάποιο δρόμο αρκετά φαρδί και χωρίς κίνηση. Στις Βρυξέλλες, επομένως, είναι χαμένο από χέρι ένα τέτοιο αυτοκίνητο αλλά πολύ σύντομα θα έχουμε αυτοκίνητα ας πούμε, τα οποία μπορούν να ε, παρκάρουν χωρίς ε, οδηγό. Ε, είναι δυνατό αυτό, αλλά δεν μας, δεν μας επιτρέπει η συνθήκη της Βιέννης να αφήσουμε ένα αυτοκίνητο να παρκάρει από μόνο του. Ο κανονισμός λέει ότι θα πρέπει να κρατάει ο οδηγός στα τιμόνι. Χωρίς μικρόφωνο κύριε Ντελβό. Ναι, αλλά τώρα βρισκόμαστε ήδη σε δεύτερη γενιά ε, ρομπότ. Ναι, και θα υπάρξει και μια μεγαλύτερη διάδραση μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ. Και όταν θα έρθει κάποια στιγμή μια άλλη γενιά ρομπότ, ε, τότε θα φτάσουμε σε ρομπότ τα οποία θα είναι όχι απλώς πιο αυτόνομα, αλλά που θα είναι αυτόνομα τελεία αυτό που σας ζητώ εγώ είναι όχι ακριβώς να ξεχάσουμε τη μακροπρόθεσμη προοπτική, αλλά να δούμε πρώτα τι μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα, τα άμεσα επόμενα χρόνια. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα του κατά πόσον θα πρέπει να δώσουμε μια νομική υπόσταση στα ρομπότ έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα, καταγράψουμε κτλ και κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικό μας σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που βασίζεται στην χρηματοδότηση, στην φορολόγηση συγγνώμη, της εργασίας, ε, όντως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το κενό που θα προκληθεί. Αυτά ήθελα να σας πω. Χαίρομαι πάντως ε, γιατί ε, διαπιστώνω ότι συμμερίζεστε κάπως τον ενθουσιασμό μου για το θέμα αυτό. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Θέλετε εν συντομία να μας πείτε τι έγινε στο, ε, στην Ουάσιγκτον. Uh, I Σας ευχαριστώ πολύ. Το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και εστίασε κυρίως σε δύο θέματα. Καταρχάς τις διαπραγματεύσεις της συμφωνίας TTIP που συνεχίζονται και έπειτα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όσο για την TTIP η εντύπωση που αποκόμισα ήταν ότι οι διαπραγματεύσεις είναι ακόμα σε ε, αρχικό στάδιο. Η νομοθεσία χρειάζεται ακόμα πολύ περισσότερες πληροφορίες, χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά. Ε, είχαμε περιορισμένη επιτυχία σχετικά στην έβρεση κάποιου με τον οποίο να διαπραγματευτούμε για την πρόταση ειδικά για το ISDS. Πιστεύω λοιπόν ότι δεδομένου ότι η πρόταση ήταν πάρα πολύ νέα εκείνη τη δεδομένη στιγμή, η ενημέρωση των μελών του Κογκρέσου σχετικά με το ISDS ήταν ε, ελλειπής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, αλλάξουμε και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Επίσης, ο, συναντηθήκαμε με έναν εμπειρογνώμονα σχετικά με τους ε, εμπορικούς αντιπροσώπους των ΗΠΑ και μας έκανα μία παρουσίαση των ελήψεων της, ε, του σήματος γεωγραφικής ένδειξης. Μας έδωσε μερικά στοιχεία και ήταν πολύ δύσκολο να συζητήσουμε και να αντιδράσουμε σε αυτά χωρίς πρώτερη ενημέρωση. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την Γραμματεία να επικοινωνήσει με τον εμπορικό εκπρόσωπο ξανά και να ζητήσει αυτά τα έγγραφα Τη παρουσίαση που μα έκανε, διότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά δεν μπορούσαμε να ε, απαντήσουμε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτά τα στοιχεία. Επίσης ε, συναντηθήκαμε με το γραφείο ε, και το γραφείο πνευματικής ε, ιδιοκτησίας και σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την μεταρρύθμιση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Βρισκόμαστε σε παρόμοιο περίπου στάδιο στις διαπραγματεύσεις και στην μεταρρύθμιση. Για παράδειγμα υπάρχουν ε, διατάξεις σχετικά με τα ε, έργα συγγραφέων, τα έργα των δημιουργών, με τα ορφανά έργα, τα έργα χωρί, που δεν μπορούν να εντοπιστεί ο δημιουργός τους, έχουμε και παρόμοιες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης. Επίσης, συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα του, της υπηρεσίας σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο δημιουργία μια υπηρεσία πνευματική ιδιοκτησία ενό τέτοιου γραφείου στην Ευρώπη. Συζητήθηκε το θέμα τη βελτίωση των συστημάτων πληροφορική. Η ανανέωση του ΟΧΙΜ η ανανέωση του συστήματος πληροφορικής εκεί σίγουρα είναι μια ευκαιρία για να συνεργαστούμε σε αυτούς τους τομείς. Επιπλέον οι Ηνωμένε Πολιτείε προσπαθούν να βελτιώσουν τα συστήματα ειδοποίησης και τα συστήματα απόσυρσης ε, πληροφοριών σε περίπτωση που ε, υπάρχουν παραβάσεις. Βέβαια προσπαθούν να αποφύγουν το ενδεχόμενο ε, λάθος Θασμένης απόσυρσης πληροφοριών. Συζητείται το θέμα των εξαιρέσεων και το ζήτημα των έργων που επανεκδίδονται. Επίσης είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το Ανώτατο Δικαστήριο και να κάνουμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων με έναν δικαστή, του δικαστή Brian, συζητήσαμε ορισμένα θέματα τα οποία είχε συζητήσει και το κοινοβούλιο, δηλαδή η προστασία ε, του, του, των public domain, τα έργα κοινή ιδιοκτησία, ανοιχτή ιδιοκτησία που πρέπει να παραμείνουν έτσι, ε, το, η νομοθεσία σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία στην Ευρώπη. Και αντίθετα με εμάς υπάρχουν σχετικά ε, λίγες πληροφορίες για πολλά θέματα τα οποία συζητούνται έντονα στην Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε. Σβιεύκα. Ευχαριστώ πολύ. Σύμφωνο 100% με αυτά που μας είπε η Τζούλια. Ε, για μια αποστολή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Από την άλλη μεριά όμως μας εξέπληξε πολύ Φανταζόμουν ότι οι Αμερικανοί εταίροι μας θα ενδιαφερόντουσαν περισσότερο και θα ήταν πιο πολύ ενημερωμένοι γιατί όταν μιλήσαμε ε, για το πώς θα έχουμε επαφές με μέλη του Κογκρέσου δεν υπήρχε τόσο ε, βαθιά γνώση. Σας τα είπε η Τζούλια για την διοίκηση και την κυβέρνηση. Σας είπε που συνδύσαμε διάφορους ε, παράγοντες. Επομένως δεν ήταν τόσο βαθιά η γνώση τους και δεν είμαι σίγουρος το κατά πόσο τα συμπεράσματά τους είναι αυτά που θα θέλαμε. Άρα θα πρέπει να δούμε κατά πόσον οι δικοί μας, ε, οι δικοί με τη σειρά τους, ξέρουν για την Αμερική. Ας πούμε γεωγραφική προστασία, ε, όπου είχαμε μια 40 λεπτή ομιλία να ε, παρουσιαστεί αλλά τα συμπεράσματα ήταν όλος διαφορετικά σε σχέση με όσα συζητούμε εδώ. Άρα, οπωσδήποτε χαρινά μου, θα χρειαστεί να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ του Κογκρέσου και του Κοινοβουλίου. Και ξέρω ότι έχουν προγραμματίσει επίσκεψη οι Αμερικανοί εταίροι μας. Επίσκεψη εδώ. Επίσης είχα την εντύπωση ότι στο Καπιτολίο δεν ενδιαφέρονταν και τόσο πολύ για το TTIP. Απασχόλησε βέβαια στην κυβέρνηση. Αλλά τελικά το κοινοβούλιο, το, συγγνώμη, το, το, το, ε, το κοινοβούλιο στο Καπιτόλιο θα αποφασίσει, το Κογκρέσο. Και όσον αφορά το copyright ήταν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ή συζητήσει. Και είδα ότι και δύο πλευρές επιδιώκουν το να βρεθούν κάποιε λύσεις είναι διαφορετικό το αμερικανικό σύστημα και δεν είναι καν ομοιογενή η ρύθμιση σε όλες τις πολιτείε. Κάθε πολιτεία έχει τη δική της ε, νομοθεσία. Πρέπει να είναι διαρκή συνταλλαγή πληροφοριών τους ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε κάποια προβλήματα τα οποία αναφύουν ή στο μέλλον όταν έρθει η ώρα των προτεραιοτητα για το TTIP. Πολύ ενδιαφέρουσα και απαραίτητη ήταν η αποστολή αυτή. Κρίμα που δεν έχουμε πιο συχνά την ευκαιρία να ταξιδέψουμε εκεί. το πιο σημαντικό μας εταίρο και εμείς θα πρέπει να θεωρούμε σημαντική αυτή τη ΣΥΠΑ. Ε, που έχουμε βέβαια τόση μεγάλη πολυμορφία και εμείς που τόσο πολύ τονίζεται φαντάζομαι ότι είναι επιφυλακτικοί για να συνεργαστούν μαζί μας. Θέλουν να γίνουν πιο στενή συνεργασία. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε που είμαστε υποταθά και πάμε τώρα εις 26 της σημερινής διατάξεως. Δηλαδή, πρόκειται για κάποια αποστολή που έκανα εγώ με την κυρία Ρέντα. Οι δυο μας. Κύριε Ρέντα, αν θέλετε μπορείτε εσείς να ξεκινήσετε. Οι κυρίες προηγούνται. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσω εγώ. Ευχαριστώ. Το παρατηρητήριο ε, παρουσίασε το πρόγραμμα εργασία από το 2016 και έκανε μια ε, συλλογή από προτάσεις ε, των Ευρωβουλευτών. Η, Ευρωπή, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έχει την άποψη ότι το παρατηρητήριο θα κάνει μια έρευνα για τα εμπορικά μυστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι μια βάση για τις συζητήσεις μας πάνω στην οδηγία για τα εμπορικά μυστικά. Θα εντοπίσουμε με τον τρόπο αυτό κάποια προβλήματα που ε, υπάρχουν σχετικά με αυτό σε διάφορα κράτη-μέλη. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε μια σύσταση για την προστασία των ε, δημόσιων ε, χώρων, των public domains, διαδικτυακών χώρων, εξετάζει την προστιθέμενη αξία των ε, χωρών αυτών σε ορισμένους τομείς πολιτισμικούς και επίσης υπάρχει και ένα άλλος πολύ ενδιαφέρον ε, τομέα στο πρόγραμμα εργασίας, οι διαφορετικά προσεγγίσεις ε, της εθελοντικής καταγραφής έργων πνευματικής ιδιοκτησίας. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, υπάρχει το σύστημα Σολιού, το οποίο προσφέρει βελτιωμένες δυνατότητες σε περίπτωση ε, δικαστικής ε, προσφυγής για κάποιο έργο. Υπάρχει επίσης ε, μεγάλη δυνατότητα χρησιμοποίησης του για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Τώρα, τα δημόσια μητρώα ήταν επίσης ένα θέμα που συζητήθηκε. Όπως ξέρετε, πέρυσι εγκρίθηκε η οδηγία για τα ορφανά έργα και η παρουσίαση του ε, μητρώου αυτού καταγραφής των ορφανών έργων ήταν ε, κάτι το πολύ θετικό. Έχουμε μέχρι τώρα περίπου 1.300 καταγεγραμμένα έργα ως όρφανα έργα, ωστόσο η πλειοψηφία τους, περίπου 750 δηλαδή, προέρχονται από ε, ένα μόνο αρχείο, το ε, Ολλανδικό Αρχείο Κινηματογράφου. Είναι λοιπόν σχετικά εύκολα τα πράγματα σε κάποιους τομείς, αλλά πάρα πολύ δύσκολα έως ε, ανέφικτα σε άλλους. από ό,τι φαίνεται, το κόστος της ε, έρευνας ε, για τους κατόχους ε, πνευματικών δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ δυσβάσταχτο για πάρα πολλά αρχεία και πολλές δημόσιες βιβλιοθήκες. Γι' αυτό λοιπόν η οδηγία για τα ορφανά έργα δεν μπορεί να εφαρμοστεί Υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες. Επίσης υπάρχουν ορισμένα έργα όπως φωτογραφίες οι οποίες δεν καλύπτονται καν από την οδηγία για τα όρφανα έργα και θα πρέπει να εξεταστεί στην ε, μεταρρύθμιση της ανομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ε, εμπορικών σημάτων. Επίσης, χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τις ε, αποζημιώσεις σχετικά με την αντιγραφή πνευματικής ιδιοκτησίας, την κλοπή πνευματικής ε, ιδιοκτησίας. Ελπίζω να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτό στο μέλλον, αλλά πέραν αυτού είχαμε και διάφορες ε, συζητήσεις που θα τις ακούσετε με περισσότερες λεπτομέρειες και από τον κύριο Κάβαντας. Ε, μία στην οποία συμμετείχα είχε να κάνει με την προστασία των καταναλωτών, μία άλλη σχετικά με την νεότητα, με τους νέους και συζητήθηκαν αρκετά θέματα τα οποία υπάρχονται στο πλαίσιο της ψηφιακής ενίας αγοράς, τα οποία έχουμε συζητήσει και σε αυτό το κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συμπληρώσω κάποια πράγματα πάνω σε αυτά που είπατε για το παρατηρητήριο, φαντάζομαι γνωρίζετε τι είναι. Πρόκειται για το ε, παρατηρητήριο ή γραφείο εναρμόνισης ιστορικής αγοράς, ε, δυναμισμός, διακρίνει αυτή την υπηρεσία ε, και γίνονται με μελέτες. Είναι σοβαρή αυτή η υπηρεσία. Υπάρχει πνεύμα επίσης αμεροληψίας, ουδετερότητος, Επομένως, για να το πούμε ξεκάθαρα, είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο. Μας παρουσίασαν αναλύσεις, μελέτες που έγιναν ε, κατά διάρκεια του χρόνου. Είναι για τα θέματα που αναφέρατε. Βεβαίω και η νέα γενιά έχει την ε, ε, ψηφιακή τεχνολογία, είναι και θέμα της ε, πνευματικής διοκτησίας και αυτό πολύ σημαντικό. Όλα όσα έχουν μιλήσει ήταν εμπεριστατωμένα. Και επομένω ήταν πολύ ενδιαφέρουσε οι ανταλλαγέ απόψεων ακριβώ γιατί όλα θα στηριζόντουσαν όχι σε συναισθηματική φόρτιση και σε ιδεολογική φόρτιση, αλλά στη λογική και ανάμεσα σε όλα τα άλλα που μας εξήγησαν μας είπαν για κάποια έρευνα του παρατηρητηρίου που έχει σχέση με την υπηρεσία αυτή για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό το λοιπόμενος λοιπόν ε, ήταν πάρα πολύ εύστοχο. Ακριβώς την ώρα των διαπραγματεύσεων για την οδηγία και το κοινοβούλιο ήθελε ένα ισορροπό κείμενο όπως και ψηφίστηκε και σας ε, πω ότι θέλω πάρα πολύ να υπάρχει ανεξαρτησία, να υπάρχει εμπιστοσύνη, εμπιστευτικότητα ε, των ε, πηγών. Και έτσι μπορούν να κάνουν το λειτουργήμά τους δημοσιογράφοι και να ενημερώνουν τον κόσμο. Όλα αυτά επομένως ε, χαρακτηρίζουν τον οργανισμό αυτό που επισκεφτήκαμε και στο τέλος επίσκεψης ή πρότεινα να δημιουργηθεί ένα ταμείο. Το ταμείο αυτό να βοηθήσει στην πρόληψη της παραβιάσεως των δικαιωμάτων μοναδικής ιδιοκτησίας. Να εμπλακούν τα κράτη-μέλη, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και μεγάλες εμπορικές εταιρείες που βέβαια έχουν μεγάλο συμφέρον, ούτως ώστε να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους για την παραγωγή τους. Οπότε να έχουμε έτσι το και δημοσίου τομέα, να δούμε τι θα γίνει. Ε, βέβαια υπάρχει και θέμα εναρμόνισης κυρώσεων και εξυγχρονισμός κανόνων λειτουργίας και να αφορά αυτό τους ενδιαμέσους θα συνεχιστεί η επαφή μας επομένως με το παρατηρητήριο όλα αυτά τα θέματα θα τα προωθήσουμε είναι θέμα οικονομικό είναι θέμα ανατικής ιδιοκτησίας βασικό θέμα για την έρευνα αλλά για την ανταγωνιστικότητα. Γιατί έχουμε 50% των εταιρεών στην Ευρώπη που χρησιμοποιούν και, με, και, και επικαλούνται τους κανόνες και όπως είπε η κυρία Ρέντα για όλα αυτά είπατε ότι ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε και ό,τι θέλετε απευθυνθείτε σε εμά και διαμέσου εμών να ενημερωθείτε. Έχουμε άλλο ένα θέμα τώρα. Ρομπέρ. Το σημείο 17 έχει να κάνει με την επικουρικότητα. Είναι συνηθισμένο υπάρχει μια διαλογημένη γνώμη που έχουμε ζητήσει από διαφορετική κοινοβούλια. Επόμενη στο Στρασβούργο, 14 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. και μετά η κανονική μας 11 Ιανουαρίου. Δευτέρα απόγευμα στις 3 φαντάζομαι. Ναι, στο Στρασβούργο θα έχουμε τη Δευτέρα μια συνεδρίαση, 14 Δεκεμβρίου. Από τις 9 μέχρι τις 10. Να έχετε πάρει και σαντουιτσάκια. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ευχάριστη συνεργασία. Καλό σας απόγευμα.